δική του, τις δικές του παρατηρήσεις. Όπως ξέρετε, ήμουν, ήμουν εδώ πριν από ένα χρόνο και η Επιτροπή σας ε, έδωσε το, ε, την δυνατότητα στην νομική υπηρεσία να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ για αυτό. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ζήτημα και πέραν όλων των άλλων για το κράτος δικαίου και την ε, εφαρμογή αυτού κυρίως ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια της χάρτας. Το πιο σημαντικό ίσως να αναφέρουμε για αυτή την απόφαση είναι ότι ε, εδρεώνει το ότι η χάρτα πρέπει πάντα να την χάνει σεβασμού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ανεξάρτητα από την απόφαση ή από το κείμενο που πρέπει να τύχει η ερμηνεία είτε είναι οδηγία που, το έχει, που την έχουν υιοθετήσει οι νομοθέτες ή είναι μια απόφαση της Κομισιόν. Η χάρτα πρέπει πάντα να εφαρμόζεται. Και αυτό είναι αυτό το οποίο έκανε και το δικαστήριο και το οποίο το οδήγησε τελικά σε αυτό το αποτέλεσμα ότι το safe harbor δεν ισχύει το βασικό μας βεβαίως καθήκον στην ε, νομική υπηρεσία είναι να υπεραμεινθούμε τη ισχύω της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων. Το βασικό μας επιχείρημα ήταν ότι η οδηγία πρέπει να ερμηνευθεί στα πλε... Ε, ε, από κοινού με τη χάρτα και όλα τα υπόλοιπα πορεύουν από αυτό. Το, το δικαστήριο ακολούθησε ακριβώς αυτή τη γραμμή και επιβεβαίωσε ότι η οδηγία είναι απολύτω σύμφωνη με τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για το λόγο αυτό το δικαστήριο δεν αμφισβήτησε κατά κανέναν τρόπο την ισχύ τη οδηγία. Αυτό είναι σαφέ. Η οδηγία μάλιστα προωθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Επομένω, όλε οι διατάξει τη οδηγία θα πρέπει να ε, ερμηνεύονται υπό αυτό το φω. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό έβριμα. Αλλά πέραν τη ερμηνεία τη οδηγία αποκινούμε τη χάρτα. Όπω είπε και το δικαστήριο, η απόφαση τη Safe Harbor τη Κομισιόν είναι ε, άκυρη. Γιατί η απόφαση αυτή δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις ε, διατάξει της οδηγίας ή τη χάρτα. Αυτά έτσι εν συντομία, εισαγωγικά. Και να πω επίσης ε, ε, το προφανές. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε γιατί ακριβώς ένας πολίτης ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Να υποβάλει ένα, μια καταγγελία σε μια εθνική αρχή. Όταν η εθνική αρχή αρνήθηκε να διερευνήσει το αίτημά του, ο, το άτομο αυτό, ο κύριος Σρέμς, πήγε στο αρώτο δικαστήριο της Ιρλανδίας. Ο δικαστής, ο Ιρλανδός δικαστής ήταν αυτός που παρέπεμψε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όπως ξέρετε, οι δικαστές, ε, οι πρωτοδίκες δεν, ε, δεν τους ζητείτε να βγάλουν απόφαση, αλλά ο κύριος, ε, ο δικαστής Χόγκαν αποφάσισε ότι αυτό ήταν ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ζήτησε απάντηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά βεβαίως πραγματικά το, ε, το μπράβο πρέπει να πάει και στον κύριο Σρέμς που το παρακολούθησε που το ε, προώθησε και στον ε, Ιρλανδό δικαστή, τον δικαστή ε, Χόγκαν, ο οποίος έστειλε την, την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και εμέσως η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων δεν προστάτευσαν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και υπό αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, αισθάνθηκε υποχρεωμένο να παρέμβει σε αυτή την υπόθεση και να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί είναι το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσει ότι η χάρτα την χάνει πλήρου σεβασμού. Και αυτό βεβαίω εξηγεί γιατί τελικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, θεώρησε την απόφαση Safe Harbor άκυρη. Ακόμη και αν ο Ριονδός, ε, μάλλον παρόλο που ο Ριονδός δικαστή, δικαστής δεν ζήτησε απόφαση επί της ε, εγκυρότητας ή όχι της απόφασης. Το θέμα ήταν, αυτό που ζήτησε ο Ριονδός δικαστής ήταν ένα θέμα ερμηνεία. αλλά όπως ξέρετε, από τις συζητήσεις μας πριν από ένα χρόνο, ήταν σαφές ότι αυτό το θέμα της ερμηνείας προφανώς ε, δημιουργεί και άλλα θέματα εγκυρότητας. Μπορεί να υπήρχε θέμα εγκυρότητας οδηγίας, το οποίο βεβαίως δεν προέκυψε, αλλά υπήρχε θέμα εγκυρότητας τη απόφαση Safe Harbor. Και αυτό ακριβώς ήταν που οδήγησε το δικαστήριο σε αυτή την απόφαση. Επίσης, ε, το ερώτημα μετά την απόφαση του δικαστηρίου είναι ποιο είναι το επίπεδο προστασίας τελικά που πρέπει να εξασφαλίζεται στα πλαίσια της χάρτας. Εδώ το δικαστήριο είναι απολύτως σαφές. Πρέπει να υπάρξει υψηλό επίπεδο προστασίας που απορρέει και από την οδηγία η οποία προβλέπει υψηλό επίπεδο προστασίας και από τη χάρτα. Οπότε το δικαστήριο επιμένει καταρχά εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και πέραν αυτού, όταν υπάρχει μεταφορά δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτη χώρα, η τρίτη χώρα θα πρέπει επίση να εξασφαλίσει την ύπαρξη υψηλού επίπεδου προστασία των δεδομένων. Το δικαστήριο εξηγεί ότι οι τρίτε χώρε δεν μπορεί να πρέπει να υποδεικνύουν το ίδιο επίπεδο προστασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τρίτε χώρε δικαιούνται να έχουν διαφορετικά μέσα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Αλλά το δικαστήριο εξηγεί ότι για να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, το επίπεδο προστασίας της τρίτης χώρας πρέπει να είναι ισοδύναμο. Όχι ισότιμο, ε, ίδιο, αλλά ισοδύναμο με το επίπεδο της προστασίας των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, το που επίσης το ξεκαθάρισε το δικαστήριο και ήταν σημαντικό για την απόφασή του, είναι ότι το επίπεδο προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται από το νομικό σύστημα της τρίτης χώρας. Και το ξεκαθαρίζει αυτό το δικαστήριο γιατί το Safe Harbor και το σχετικό σύστημα είναι σύστημα αυτοπιστοποίησης, δηλαδή ένα σύστημα εθελούσιο για τις ιδιωτικές εταιρείε. Αν μια ιδιωτική εταιρεία ε, ενταχθεί σε αυτές τις αρχές, αυτές οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, απέναντι σε αυτή την εταιρεία. Αλλά οι αρχέ των ΙΠΑ ε, δεν δεσμεύονται από αυτές τι αρχέ του Safe Harbor. Το νομικό σύστημα δεν υπόκειται σε αυτή τη, σε αυτή τη συμφωνία του Safe Harbor. Είναι ε, οι εταιρείε ιδιωτικέ μόνο που εντάσσονται. Οπότε το δικαστήριο Γι' αυτό ακριβώ θεώρησε ότι πρέπει η απόφαση αυτή να θεωρηθεί άκυρη. Γιατί η Κομισιόν στην απόφαση Safe Harbor δεν λέει ότι η ΕΠΑ και το νομικό σύστημα των ΕΠΑ προσφέρει επαρκέ ή ισότιμο επίπεδο προστασία. Λέει ότι απλώ οι αρχέ αυτέ δεσμεύουν τι ιδιωτικέ εταιρείε. Οπότε κατά μία έννοια, και σε αυτό καταλήγει το δικαστήριο, η απόφαση Safe Harbor της Κομισιόν ουσιαστικά ε, είναι τελείως εκτός θέματος. Δεν, αφο, δεν ασχολείται με το βασικό ζήτημα που απορρέει από την οδηγία και που είναι να δηλώσει η Κομισιόν ότι η νομοθεσία και το νομικό σύστημα της τρίτης χώρας εξασφαλίζει το υψηλό επίπεδο προστασίας. όλα αυτά το δικαστήριο δεν έμεινε σε αυτό, πήγε λίγο παραπέρα και εξήγησε λεπτομερέστερα το τι γίνεται σε περίπτωση που η νομοθεσία της τρίτης χώρας προβλέπει ε, κάτι που ε, αντίκειται στην ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία και πώς αυτό μπορεί να διολογηθεί. Το δικαστήριο εδώ εφαρμόζει το ίδιο που έκανε και πριν στην, στην απόφαση της Ιρλανδίας για τα ψηφιακά δικαιώματα. Και εκεί υπήρχε ε, θέμα για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία υιοθετεί ένα μέτρο το οποίο, ε, δεν, ε, το οποίο αντίκειται στα θεμελιώδη δικαιώματα. Και το δικαστήριο είπε και επέμεινε στις απαιτήσει της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Και αυτό που έκανε τώρα το δικαστήριο για τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων είναι να χρησιμοποιήσει ακριβώς την ίδια λογική για τη νομοθεσία της τρίτης χώρας. Οπότε, μια τρίτη χώρα για να μπορεί να παράσχει νομικά το ίδιο επίπεδο προστασίας θα πρέπει αυτή η νομοθεσία να είναι αναλογική και απαραίτητη και ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο το δικαστήριο αφηρημένα μεν αλλά το εξηγεί δε ότι σε καμία περίπτωση στην Ευρώπη καμία νομοθεσία δεν θα μπορούσε είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να παράσχει μαζική παρακολούθηση. Το δικαστήριο ε, ε, χρησιμοποιεί πολύ σαφή ορισμό δεν λέει ε, μαζική παρακολούθηση, ο Γενικός Αγγελέας το λέει, αλλά εξηγεί ακριβώς τι σημαίνει. Σημαίνει πρόσβαση σε γενική ε, κλίμακα στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επικοινωνιών όλων των ατόμων. Ουσιαστικά μαζική παρακολούθηση. Οι αρχές δηλαδή μπορούν να διαβάσουν όλα τα email όλων των πολιτών όποτε το επιθυμούν. Τι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο είναι αδύνατο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετηθεί τέτοια νομοθεσία που θα επιτρέπει αυτό. Οπότε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται αυτό. Αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μια χώρα παρέχει ε, τέτοιο επίπεδο υψηλό προστασία εφόσον στην νομοθεσία τη υπάρχει διάταξη που επιτρέπει τη μαζική παρακολούθηση ή αυτό που ορίζει το δικαστήριο στη μαζική παρακολούθηση. Δεύτερο, ε, δεύτερη σημαντική ε, αρχή είναι ότι η νομοθεσία δεν προβλέπει ένδικα μέσα. Και όταν δεν προβλέπει ένδικα μέσα, σημαίνει παραβίαση των, των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί στο άρθρο 47 τη Χάρτα αναφέρονται σαφώ τα ένδικα μέσα. Αν η νομοθεσία δεν προβλέπει ένδικα μέσα για, την, για τους Ευρωπαίους πολίτες, ουσιαστικά δεν, ε, δεν ε, στέκεται στο ύψος του επίπεδου προστασίας που θέλει να παράσχει. Και για τις τρεις αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε λοιπόν ε, πρόβλημα. Όχι, αυτό, όχι του ότι ξεπερνούσαν αυτό που ήταν απαραίτητο και ανάλογο, αλλά όπως είπε και ο Γενικός Αγγελέας ε, ήταν εξαιρετικά σημαντικό και πρώτη φορά το δικαστήριο βλέπει μια υπόθεση όπου η ουσία, η ουσία ενός, ε, ενός ε, θεμελιώδους δικαιώματος καταπατείται. Το θεμελιώδους δικαιώματος δηλαδή της προστασίας της ιδιωτικότητας. Ε, ε, στην, ε, στην, στην οδηγία για την ε, διατήρηση των δεδομένων δεν ήταν το ίδιο βέβαια. Εκεί μιλούσαμε για μεταδεδομένα. Δεν μιλούσαμε για, τα, για, την, για το τι διαβάζουν και αν διαβάζουν το περιεχόμενο των email οι αρχέ. Αλλά τώρα, σε τούτη την περίπτωση, η NSA, η υπηρεσία της των ΗΠΑ, μπορεί να διαβάσει όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες των πολιτών. Και αυτό βεβαίως δεν είναι, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό στα πλαίσια της χάρτας και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Υπήρχε και άλλη μια πτυχή σε αυτή την υπόθεση, όχι κατά ανάγκη ε, σχετιζόμενη με την ε, εγκυρότητα, αλλά το δικαστήριο ε, ερμήνευσε τις διατάξεις της τρέχουσας οδηγία για την προστασία των δεδομένων και εκεί κατέστησε σαφές ότι αυτό πρέπει να ερμηνευθεί ως διάταξη που επιτρέπει στις αρχές προστασίας των δεδομένων των, κρατών μελών να ελέγχουν την, μεταφορά, την ανταλλαγή αυτή των δεδομένων. Και επίσης κάνει μια σημαντική προσθήκη ενδιαφέρουσα το δικαστήριο και λέει ότι αυτό που πρέπει να γίνει σε μια περίπτωση όπου μια εθνική αρχή προσθέτει δεδομένων διερευνά το ζήτημα και βλέπει ότι όντως η μεταφορά αυτή των δεδομένων παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τότε, λέει το δικαστήριο, η αρχή προσθέτει δεδομένων πρέπει να ε, πάει στο Εθνικό Δικαστήριο και να ζητήσει από το Εθνικό Δικαστήριο να βγάλει μια, πρωτό, μια απόφαση. Οπότε ο δικαστής μπορεί να ακυρώσει ουσιαστικά ή να θεωρήσει ως άκυρη ή μη ισχύουσα την απόφαση της Κομισιόν. Οπότε το δικαστήριο τώρα δημιουργεί ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι αρχές των κρατών μελών μπορούν να πάνε στο εθνικό τους δικαστήριο και από εκεί και πέρα το δικαστήριο να, κάνει, να λάβει αυτή την απόφαση. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τη νομική του πλευρά. Οπότε, σε ό,τι αφορά την ε, νομική έτσι, αρχιτεκτονική στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως για τα θεμελιώδη δικαιώματα, πραγματικά αυτή η απόφαση έχει πολύ σημαντικές συνέπειες. Θα σταματήσω εδώ. Βεβαίως, αν υπάρχουν ερωτήματα, ευχαριστώ να σας απαντήσω. Ε, Thank you very much. Ευχαριστώ, κύριε Ρέη. ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις σας μία ερώτηση για τις επιπτώσεις αυτής της ε, απόφασης για τη μαζική παρακολούθηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε ότι το δικαστήριο φρονεί ότι καμία νομοθεσία που να αφορά την μαζική παρακολούθηση δεν μπορεί να ισχύσει στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Υπάρχει όμως τέτοιου είδους ε, νομοθεσία. Αν το Facebook έχει ε, κέντρα δεδομένων στην Σουηδία. Οι ιδιοκτικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα εκεί και μπορεί κάποιος πολίτης μέσω της Εθνικής Αρχής ε, Προστασίας Δεδομένων ε, να προσβάλλει το κέντρο το οποίο μπορεί να δώσει σε μια άλλη χώρα τα δεδομένα του σε κάποιον τρίτο. Είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα. Βασικά πρέπει να πω ναι. Τώρα είχαμε να κάνουμε με μεταφορά στοιχείων σε διεθνές επίπεδο. Τώρα για νομοθεσία τρίτων κρατών. Αλλά είναι δυνατόν και λέει το δικαστήριο ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν θα έπρεπε να επιτρέπει δεδομένου ότι υπάρχει η χάρτα προστασίας των, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύει η κοινοτική νομοθεσία να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά την ε, ηλεκτρονική επικοινωνία, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ως σημείο κίνηση ότι ο κοινοτικό νόμος, η κοινοτική νομοθεσία ισχύει. Αλλά θα πρέπει κατά περίπτωση να εξετάσουμε περί τίνος πρόκειται, διότι και εδώ ίσως θα έχουμε επιπτώσεις με διάφορα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται εντός των κρατών μελών με διαφορετικό τρόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Άντερσον. Και εγώ σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο πράγμα που ερώτησε και η Τζούλια. Θα δούμε κατά της, ε, των Σουηδών για τα θέματα αυτά της ε, επικοινωνίας και της ε, διαβίβασής τους ε, να γύρονται πολλά θέματα. Μου αρέσει λοιπόν αυτή η υπόθεση γιατί έχει συνέχεια. Ο κύριος Μαρίνιο Πίντο. Η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι εξαιρετικά σημαντική. Ακόμη ίσως δεν μπορούμε να, τη, να δούμε πόσοι σημασία μπορεί να έχει στο άμεσο μέλλον για την προστασία της προσωπικής ζωής του κάθε πολίτη. Το θέμα αυτό της ιδιωτικής ζωής είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να συνοψιστεί μόνο σε αυτό που λέμε η ιδιωτικότητα της ζωής, διότι υπάρχουν ε, πάρα πολλά ε, δεδομένα τα οποία αφορούν τον κάθε πολίτη στην ε, ιδιωτική του ζωή. Τώρα, το θέμα της ιδιωτικότητας είναι κάτι το οποίο είναι ίσως ένα θέμα το οποίο δεν χρειάζεται να προστατεύεται στο έπακρο. Αλλά πρέπει να πω ότι είμαστε μπροστά σε μία διαδικασία αλλαγής των πάντων. Είναι πάρα πολύ ταχεία η εμπλοκή ε, των μοντέρνων ε, τεχνολογιών και η νομοθεσία είναι πάντα ένα βήμα πίσω. Τώρα, σε περίπτωση μιας μυστικής υπηρεσίας, κρατικής υπηρεσίας των Αμερικανών, συγκεκριμένη περίπτωση, που θέλει να ελέγχει τι κάνει ένας Πορτογάλος πολίτης που κάνει διακοπές ε, στην Ιαπωνία βάσεις, με, χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων που βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα δημιουργεί. Έχουμε τέσσερις νομοθεσίες, τέσσερις χώρες και πώς μπορούμε να διευκρινίσουμε τα πράγματα, δούμε τι ισχύει για ποιον. Πιστεύω λοιπόν ότι Αυτό το θέμα που άπτεται του θέματος που συζητούμε είναι το επίπεδο προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων θα πρέπει να είναι δύναμο με αυτό που χρησιμοποιούν τα κράτη όταν πρόκειται για έκδοση ενός ε, πολίτη. Η δική μας νομοθεσία απαγορεύει την έκδοση ενός Πορτογάλου πολίτη σε άλλη χώρα όταν ε, τίθεται θέμα ισόβιας κάθεξης ή θανατικής ποινής. Και λέει ότι δεν μπορεί σε αυτή την περίπτωση να εφαρμοστεί σε μια άλλη χώρα αυτού του είδους η ε, κύρωση, αν θέλετε. Και ποια είναι εδώ η δευτερεύουσα ιδέα. Δεν αρκεί μια δήλωση των αρχών της χώρας που έχει τα δεδομένα και που λέει ότι θα τα προστατεύσει και δεν θα τα χρησιμοποιήσει για χύψη ψ, σκοπούς. Και καμία νομοθεσία δεν δίνει τέτοιου είδους εγγύηση. Άρα το διατάφτα είναι ότι εάν οι πολίτες παρακολουθούν ε, συνεχώς ε, τα κοινοβούλια τα δικαστήρια, τα δικαιοδοτικά ε, μέσα συνέχεια παρακολουθούν πώς προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα και επισημαίνουν τι γίνεται, μόνον έτσι θα μπορέσει κανείς να πιστεύει ότι προστατεύεται. Χαιρετίζω λοιπόν το ότι χρειάστηκε να ασχοληθούμε με αυτή την υπόθεση για να κάνουμε τις παρατηρήσεις αυτές που είναι τόσο σημαντικές. Ο κύριος Καστέ. Και εγώ χαίρομαι που υπήρξε αυτή η απόφαση γιατί αυτό δείχνει ότι το δικαστήριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. θα μπορούσαμε να ρωτηθούμε τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής στην πρακτική ζωή. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά δεδομένων από την Ευρώπη στις Ηνωμένε Πολιτείε. Τι σημαίνει αυτό, ότι το Facebook και το Google θα μπορούσαν να συνεχίσουν να συμπεριφέρονται όπως έκαναν μέχρι τώρα και τι μέσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να κάνει κανείς κάτι σε ό,τι αφορά αυτή την απόφαση. κυρία Χάουταλα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι πραγματικά είναι μία πολύ σημαντική απόφαση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων με τις νομικές υπηρεσίες το θέμα είναι να δούμε ποιε είναι επιπτώσει. Έγιναν ορισμένε προτάσει, υποδείξει σχετικά με το ποιε θα μπορούσαν να, είναι οι επιπτώσει. Παρατέθηκε για το παράδειγμα τη Σουηδία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις σε επίπεδο μεταφοράς δεδομένων και τη συμφωνία μας με άλλες τρίτες χώρες, για παράδειγμα τη Ρωσία. Το θέμα είναι πώς μεταφέρονται τα δεδομένα σε μια χώρα σαν την Ρωσία. Πιστεύω ότι αυτό θέτει κάποιο ερώτημα σε ό,τι αφορά την παράνομη φύση των ε, υπηρεσιών πληροφοριών. Στο παρελθόν οργανώθηκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση για τις υπηρεσίες πληροφοριών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με αυτό που συζητάμε. Υπάρχουν φορείς στην, στις χώρες μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι δεν πιστεύουν στα ίδια δικαιώματα όπως ε, άλλοι φορείς. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια έτσι ώστε να μην καταφεύγουν στα άκρα. Τέλος, γνωρίζουμε ότι οι αρχές προστασίας των δεδομένων από τις 28 χώρες μέλη το συζητάνε αυτό το θέμα μεταξύ τους. Ενδεχομένως, κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση που έχουμε κάποια αρμοδιότητα να συνεχίσουμε τη συζήτηση, μήπως θα πρέπει να συζητήσουμε με τον επόπτη για την προστασία των δεδομένων. Για να δούμε ποιε είναι οι επιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να ευχαριστήσω τις νομικές υπηρεσίες για την σαφή εξήγηση που έδωσαν σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις που θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φεράρα. Mm. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πω είμαι υπέρ της τελευταίας αυτής απόφασης γιατί είναι μία απόφαση ότι η χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί ποτέ να τίθεται υποσυζήτηση. Πραγματικά όμως αναρωτιέμαι και θα ήθελα να διατυπώσω άμεσα ένα ερώτημα Ποιες είναι οι πρακτικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτή η απόφαση στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Τι επιπτώσεις θα μπορούσαν να προκύψουν για το TTIP. κύριος Λεμπουχατό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2015 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι θετική διότι προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και μας προστατεύει κατά της πολύ ταχείας διαβίβασης προσωπικών δεδομένων. Έχει όμως και κάποια ανισχυτικά σημεία διότι ε, μας δείχνει με ποιο τρόπο ομό φέρεται ώρες ώρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να επισημάνω δύο ε, θέματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει υπερβολική εξουσία εκ μέρους της Επιτροπής, διότι μειώνει τα δικαιώματα όπως στη δική μας περίπτωση της ΚΝΙΛ. Δηλαδή, είναι ανισχυτικό ότι ξεπερνάει τα όρια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι το διαπιστώνει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεύτερον, το δικαστήριο κατά κάποιο τρόπο ε, είναι κατά του υπερβολικού, της υπερβολικής αισιοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέγει ότι το επίπεδο προστασίας των δεδομένων εδώ είναι το ίδιο με τη ΣΥΠΑ. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ανησυχητικό σαν αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κυρίως αυτών που περνάνε μέσω του Facebook, διότι βλέπουμε ότι τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά στο Facebook, χωρίς καμία προστασία, διαβιβάζονται στη ΣΥΠΑ. Εμένα με ανησυχεί πολύ αυτό και θα ήθελα να ε, ε γενικεύσω το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι δεν εμπιστεύομαι πολύ την Επιτροπή και ό,τι διαβάζω με ανησυχεί. Νομίζω ότι σε θέματα τέτοιου είδους γενικευμένης κατασκοπίας τον είπα προς τις χώρες όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Δεν λέω ότι δεν είναι εταίρος μας, αλλά πρέπει να διαπιστώσω ότι δεν συμπεριφέρεται σωστά τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζεται λοιπόν να έχουμε τέτοια υπερβολική ασιοδοξία. Και με ανησυχεί το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τις διαπραγματεύσεις για το TTIP που είναι μια συνθήκη κατά της οποίας εγώ είμαι κάθετα αντίθετος και διαπιστώνω ότι είμαστε πάλι σε κατάσταση πλήρους αισιοδοξίας όσον αφορά ότι γίνεται με τη ΣΥΠΑ. Έτσι θα προσπίσουμε τα συμφέροντα τα ευρωπαϊκά. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την απόφαση υπάρχουν πιο ενισχυτικά σημεία παράθετικα. Ευχαριστώ. Uh, that was the end of the list before you... Φτάσαμε στο τέλος του καταλόγου των αγοριτών. Και εγώ έχω μια ερώτηση να μας εξηγήσετε, όταν εξηγήσετε τις επιπτώσεις, πείτε μας, έχει κάποια σχέδια η Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο θα διαπραγματευτεί με τις ΕΠΑ την προστασία των δεδομένων, διότι πρέπει να πω ότι υπάρχουν τόσο πολλές αντιρρήσεις για το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις ΕΠΑ, που πιστεύω ότι πραγματικά έχουμε στο θέμα αυτό μεγάλα προβλήματα. Σας δίνω το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω ίσως όχι με την ίδια σειρά με την οποία τέθηκαν. Αρχίζω με το θέμα που αφορά την κατάσταση σε άλλες τρίτες χώρες, διότι αυτό θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε το τι πρέπει να κάνουμε τώρα με τη ΣΥΠΑ διότι είπα είναι στην ίδια ε, θέση ίσως και με άλλες χώρες, εκτός από κάποιες λίγες. Οι περισσότερες χώρες, μεγάλες χώρες, η Ινδία, η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Κίνα, κατά κάποιο τρόπο ε, δεν έχουν ε, την ε, ίδια θέση, η θέση της Κομισιόν δεν είναι επαρκής αν θέλετε, δεν τους προστατεύει και έχουν τα ίδια προβλήματα. Το άρθρο 26 της παρούσας οδηγίας ε, για την πρόταση καταλληλότητος που αφορά το θέμα αυτό, έτσι όπως συζητείτε στο άρθρο 25, επίσης ισχύει και πρέπει να πω ότι στην πρώτη περίπτωση, σε ατομικές περιπτώσεις, μπορεί κάποια ε, δεδομένα να διαβιβάζονται εάν ε, προκαλούν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, φερρυπίν για την ε, μία σύμβαση αλλά δεν αφορούν γενικευμένη διαβίβαση δεδομένων. Πάντα οι αρχές προστασίας δεδομένων μπορούν να επιτρέψουν την διαβίβαση δεδομένων όταν υπάρχει η επαρκής προστασία. Και αυτό είναι κάτι που προβλέπεται σε κάποιες συμβάσεις. Υπάρχουν λοιπόν κανόνες και έτσι μπορούν αυτή τη στιγμή να πούμε ότι γίνονται διαβιβάσεις και προς άλλες χώρες. Θα πρέπει όμως να προσθέσω ότι ό,τι είπε σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο θα ισχύει και όχι μόνο για το άρθρο 25 αλλά και για το 26. Εάν θεμελιώδη δικαιώματα και η ουσία τους τίθεται ένα αμφιβόλο, είναι πολύ δύσκολο και σχεδόν αδύνατο να δούμε πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άλλοι και να ισχύσουν άλλοι κανόνες. Το πρόγραμμα που ταυτοποίησε και εντόπισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι η νομοθεσία των ΗΠΑ που επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να κάνουν τέτοιου είδους επιτήρηση, αν θέλετε, παρακολούθηση. Και δεν έχουμε κατάλληλα μέσα προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών. Αν δεν αλλάξει η νομοθεσία λοιπόν στις ΗΠΑ, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε εμείς κάτι καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες άλλες ε, ε, νομικές δυνατότητες ανοίγονται μπροστά μας. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να πω ότι είναι πολύ πρόσφατη αυτή η απόφαση, εδώ και μία εβδομάδα και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, εφαρμογή στην πράξη όλων αυτών των αρχών που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση αυτή. Τώρα, αυτό αφορά τις τρίτες χώρες και η ΕΠΑ δεν είναι όπως κάποιες άλλες τρίτες χώρες. Και αυτό απαντά και το ποιες είναι οι επιπτώσεις θα πρέπει να εξετάσει τώρα η Κομισιόν και οι Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Πιστεύω ότι ήδη αυτή την εβδομάδα την προηγούμενη ε, συνήλθαν ε, με πήγουσες διαδικασίες όλες οι αρχές για να συζητήσουν την απόφαση αυτή και τις επιπτώσεις. Άρχισαν λοιπόν οι συζητήσεις τους και από ξέρω άρχισε και η Κομισιόν ή συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ για το TTIP και ασχολείται ε, με το θέμα αυτό. Ακόμη δεν γνωρίζει το Κοινοβούλιο ποια είναι το περιεχόμενο όλων αυτών των συζητήσεων και είναι δύσκολο στην παρούσα στιγμή να δούμε τι θα, ποια θα είναι η έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων, διότι προσπαθεί να ζητήσει την επιβολή 13 μέτρων η Κομισιό από τη ΣΥΠΑ ώστε να υπάρχει επαρκής ε, προστασία. Πιστεύω ότι γύρω στις 11, 11 από αυτά τα μέτρα έχουν συμφωνηθεί, αλλά τα δύο που είναι τα πιο σημαντικά ακόμη είναι αντικείμενο Διαπραγματεύση. δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ βασικό θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται στο στάδιο ακόμη της ε, συζήτησης και δεν ξέρουμε ποιο είναι ακόμη το διατάφτα. Το θέμα των ε, υπηρεσιών πληροφοριών είναι ένα σημαντικό θέμα. Ήδη το Κοινοβούλιο ασχολείται με τις δραστηριότητες της υπηρεσία πληροφοριών των ΙΠΑ, ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και νομίζω ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι πολύ σημαντική για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στα πλαίσια της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη ε, εξετάσει και την ομολογία που απορρέει από το ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Εν πάση περιπτώσει, συμβαδίζουν κατά κάποιο τρόπο οι προσεγγίσεις και των δύο αυτών ε, δικαστηρίων και ακόμη και με την εφαρμογή της ε, Σύμβασης του Στρασβούργου για τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εν πάση περιπτώσει λέω πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση και θα πρέπει να ασχοληθούμε περαιτέρω με την εξέτασή της ενδελεχώς. TTIP οι σχέσεις μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και διεθνών συμβάσεων. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν θα πάρουμε θέση για να πω σε σχέση με αυτή την απόφαση του δικαστηρίου τι θα συμβεί με το TTIP, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το πολύ σημαντικό και εξορισμού δεν μπορεί να υπογράψει μία σύμβαση, μία συμφωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται μέσω της χάρτας προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσουν το κατά πόσον είναι δυνατόν να ληφθούν κάποια μέρα συγχρόνως εξασφαλίζοντας την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό το θέμα το παρακολουθούμε εκ των σύνεγγες. Επίσης, ελέγχθη ότι ξεπερνά τα όρια των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα αυτό. Ίσως δεν το εξήγησα πολύ στην ε, παρατήρησή μου. Είναι ένα θέμα το οποίο φέρε επιτάπητος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας αφορά διότι θα πρέπει να δούμε σε ποιο μέτρο η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δίδει εξουσίες στην συγκεκριμένη περίπτωση σε αυτή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Safe Harbor. Είναι κάτι το οποίο ανέφερα προηγουμένως και μπορεί μόνο η Κομισιόν να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες ε, τις έχουν ε, δοθεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν δόθηκε ε, η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία να ε, ενεργήσει σε, πρώτη, σε επίπεδο διότι υπεύθυνοι για αυτές τις ε, περιπτώσεις ήταν οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων που πρέπει να έχουν και την δυνατότητα σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα η αξιώσει εκ μέρους κάποιου να κάνουν τις έρευνες και ξέρουμε ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση ξεπέρασε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ε, θεωρεί και το ίδιο το δικαστήριο ότι είναι άκυρη η απόφαση Safe Harbor. Επίση, η απόφαση λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να πάρουν αποφάσεις σε κάποια θέματα. Οπότε γι' αυτό το δικαστήριο θεώρησε ότι η πρόταση αυτή δεν είναι, είναι άκυρη γιατί δεν, α, δεν έλαβε υπόψη αυτή την οπτική. Και αυτό είναι ενδιαφέρον για το Κοινοβούλιο γιατί η Κομισιόν δρά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τη έχουν αποδοθεί και πρέπει φυσικά να τις σέβεται. Ελπίζω ότι έχω απαντήσει στα περισσότερα σημεία. Αν υπάρχουν κάτι, κάποιο, αν υπάρχει κάποιο ερώτημα που έχω ξεχάσει, παρακαλώ να μου το υπενθυμίσετε. Η κυρία Ρέντα θέλει πάλι το λόγο. Ναι. Μια έξτρα ερώτηση για αυτό που μας εξηγήσατε μόλις. Αν κατάλαβα καλά, η Κομισιόν δεν είχε την αρμοδιότητα να πάρει αυτή την απόφαση. Αυτό ισχύει και για άλλες τρίτες χώρες που έχουν ε, λάβει τέτοιες συνολικές διατάξεις. Γιατί αναφέρεται ότι υπάρχουν και 4-5 ακόμα. Και επίσης, υπάρχει κάποιος κίνδυνος να ε, πάει αυτό, να επιδεινωθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, οι εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων τι περιθώριο λιγμών έχουν μετά την απόφαση, από ό,τι καταλάβα, η Ιρλανδική Αρχή είναι αντικείμενο έρευνα στα πλαίσια αυτή τη ε, υπόθεση του κυρίου Σρέμ. Αν δηλαδή μετά την ε, έρευνα ε, βρεθεί ότι, για παράδειγμα, οι Αμερικανικέ Αρχέ έχουν τέτοιε συνολικέ δικαιοδοσίε παρακολούθηση, όπω α πούμε για τα δεδομένα στο Facebook, θα υπάρχει περίπτωση να αποφασιστεί ότι τα δικαιώματα του κυρίου Σρέμς δεν παραβιάστηκαν γιατί δεν μπορεί να δείξει ότι έχουν αναλυθεί, έχουν ε, ε, δημοσιευθεί κάποια δικά του προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή αν υπάρχει μία αρχή εθνική προσωπικής δεδομένων που αποφασίζει έτσι τι κάνουμε, όλες οι εταιρείες βάζουν ας πούμε την έδρα τους σε αυτή την ε, χώρα και μπαίνει, υπάρχει κάποιος περιορισμός, είναι δυνατόν να βάλουμε κάποιο περιορισμό σε αυτό. Και επίσης στην απάντησή σας θα μπορούσατε να μας πείτε τι γίνεται με το βάρος απόδειξης σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ναι. Ενδιαφέρουν τα ερωτήματά σας για τις ε, χώρες που ήδη έχουν τη δυνατότητα αυτή, προφανώς της αφορά. Ε, δύο λόγους έδωσε το δικαστήριο για να ε, αιτιολογήσει την ε, μη εγκυρότητα του, της απόφασης. Καταρχάς γιατί μπορεί όντως να έχουν το ίδιο επίπεδο μη εγκυρότητας και αν ε, και στις προηγούμενες ε, ε, περιπτώσεις περιορισμού των, εθνικών, των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων από την Κομισιόν στα πλαίσια του άρθρου 3 θα μπορούσε να συναχθεί ως, ως συμπέρασμα ότι η απόφαση είναι άκυρη. Ο πρώτος λόγος που έδωσε το δικαστήριο και που δεν τα πήγε καλά η Κομισιόν στα πλαίσια της απόφασης Safe Harbor ήταν ότι η Κομισιόν απέτυχε στο επίπεδο του, να, απέτυχε να ε, κατανοήσει το επίπεδο προστασία που δίνει το νομικό σύστημα των ΗΠΑ, που δεν είναι επαρκέ. Το σύστημα αυτό είναι θελοντικό για τι εταιρείε, όπω είπαμε. Ε, σε περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα στι υπόλοιπε εταιρείε ε, πρέπει να ελεγχθεί αυτό, η Κομισιόν να έχει επιβεβαιώσει ότι αυτέ οι χώρε ε, παρέχουν ένα ε, επαρκές νομικό, ένα επίπεδο προστασίας στα πλαίσια του δικού τους νομικού συστήματος μπορεί τα συμπεράσματα να είναι διαφορετικά, αλλά η λογική είναι η ίδια. Μπορεί να υπάρχουν τρίτες χώρε που να έχουν συγκεκριμένη νομοθεσία προστασία δεδομένων, η οποία να παρέασχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας, αποδεκτό από την Ένωση. Το δεύτερο ερώτημα... Α, ναι, το βάρο απόδειξη. Yes, this is an issue. Um... Ναι, αυτό. Εδώ υπάρχει κάποιο περιθώριο ελιγμόνο Είναι ανεξάρτητοι και μπορούν εξορισμού να επιλέξουν. Αυτή ήταν μια κάπως ειδική περίπτωση γιατί έρχεται στην Ιρλανδία δεν είπαν επιλέγω να μην διερευνήσω ε, είπαν ότι απέχω πολύ από το να διερευνήσω. Αυτό λοιπόν πυροδότησε αυτή την κατάσταση. Δεν υπήρχε δηλαδή ε, νομικό εμπόδιο για την έρευνα. Το αντίθετο, υπάρχει υποχρέωση έρευνας. Αλλά το θέμα είναι σε τι συμπέρασμα καταλήγουν οι αρχές μετά τη διεξαγωγή της ε, έρευνας. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την, ε, το φορέα προστασία προσωπικών δεδομένων. Αν υπάρχουν όμως ε, περιπτώσεις που επιλέγεται να μην δοθεί συνέχεια, τότε ο φορέας δεδομένων μπορεί να το υποβάλει το θέμα αυτό στο Εθνικό Δικαστήριο. Η αρχή ε, δεδομένων μπορεί να το υποβάλει στο δικαστήριο. Έχουμε να κάνουμε με μια οδηγία που ζητάει από τις χώρες μέλη να εφαρμόσουν το, εθνικό, το ε, κοινοτικό δίκαιο. Ο εθνικό, το εθνικό δίκαιο είναι εκείνο που θα καθορίσει το βάρος της απόδειξης. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισοδύναμη προστασία όταν μιλάμε για εθνικό και για νοσιακό δίκαιο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει προστασία και το ε, υποχρέωση, η απόδειξη δεν πρέπει να είναι τόσο ψηλή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, διάφορες αρχές και τις διάφορες χώρες, πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα. Είναι κάτι που είναι υποσυζήτηση στα πλαίσια της ε, μεταρρύθμισης που αφορά την προστασία των δεδομένων και υπάρχει πρόταση να υιοθετηθεί αυτός ε, ένας μηχανισμός που είναι ένας μηχανισμός για τον μελλοντικό κανονισμό. Θα έλεγα λοιπόν ότι ελπίζουμε οι λύσεις αυτές να είναι καλές για το μέλλον. Για την ώρα θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια της οδηγίας αλλά εάν χρειαστεί θα υπάρξει μία μεταρρύθμιση στο τέλος της ε, χρονιάς και θα υπάρξει μία καινούργια νομοθεσία. Και ενδεχομένως αυτή θα δώσει μια πληρέστερη απάντηση. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Uh, uh, thank you. I would... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις νομικές υπηρεσίες. Ε, δεν ζήτησε κανένας άλλος το λόγο. Από ό,τι φαίνεται εξαντλήσαμε την ημερησία διάταξη. Σας αύριο το πρωί. Ευχαριστώ.